Darf Παρακαλώ καθίστε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζουμε με την ε, σύνοδο η οποία διακόψει στις 4 Ιουλίου του 2013. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης.